Καλημέρα. Καλωσορίζω όσους είναι εδώ, ελπίζοντας ότι θα έρθουν και άλλοι. Δεν ήταν δική μας απόφαση να κάνουμε συνεδρίαση αμέσως μετά τη χθεσινή γιορτή, αλλά έχουμε και το θέμα της διερμηνίας που έχουμε Δευτέρα, Τρίτη ή Τρίτη, Τετάρτη. Εν πάση περιπτώσει, δεν είχαμε δυνατότητα να επιλέξουμε άλλη ημέρα. Γι' αυτό είμαστε και πέντε χωρίς τους συνεργάτες. Ευτυχώς που είναι και αυτοί. Αν και είμαστε λίγο... Α, έξι είμαστε τώρα. Εντάξει. Έχουμε λοιπόν σήμερα διερμηνία σε όλα εκτός από λιθουανικά, λετονικά, εστονικά, σουηδικά και μαλτέζικα. Έχουμε κροατικά για πρώτη φορά, αλλά δεν ήρθε ο συνάδελφος. Πάμε στο σημείο... Α, υπάρχουν ε, αντιρρήσεις στην ημερήσια διάταξη. Όχι. Ο κύριος Φοντάνα δεν μπορεί να έρθει σήμερα το πρωί και παρακαλεί να μεταθέσουμε το θέμα για το απόγευμα. Και πάμε στο σημείο 3 και 4 στην ημερήσια διάταξη που είναι το πρόγραμμα πλαίσιο Horizon 2020. Η Έμα Μακλάρκιν είναι η συγγήτρια που το απόγευμα δεν θα μπορεί να έρθει γιατί έχει ταξίδι. Θα δει τη Βασίλισσα. Ε, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους ως εισηγήτρια των δύο ε, θεμάτων, των γνωμοδοτήσεων και από την ε, Ήτρε που είναι επί της ουσίας, θα αναφερθώ και στα δύο. Ο στόχος είναι να συνδυάσουμε όλη τη χρηματοδότηση έρευνας και καινοτομίας σε ένα ε, πλαίσιο. Εμείς έχουμε τρία υποθέματα. Ε, χαίρομαι για την ε, ε, βοήθεια στο θέμα της αριστείας που είναι βασικό για την καλή έρευνα και για τις χρηματοδοτικές επιλογές. Επίσης χαιρετίζω το φιλόδοξο προϋπολογισμό του Horizon 2020. Ε, εδώ υπάρχει προστιθέμενη αξία και χρειάζεται υποστήριξη. Ε, έτσι λοιπόν ε, θα πρέπει να αυξηθεί ο προϋπολογισμός για αυτό το σημαντικό πρόγραμμα. Όμως, στα πλαίσια του προϋπολογισμού Horizon 2020 πρέπει να επανεστιάσουμε στις ε, δημοσιονομικές προτεραιότητες τα τρία δις πάνε για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και τεχνολογίας. Πρέπει όμως να αξιολογήσουμε την προστιθέμενη αξία για να είναι σαφές πού δαπανώνται τα χρήματα έτσι θα έχουμε μεγαλύτερη αξία στα χρήματά μας σε σχέση με άλλες προτεραιότητες το 2020, το Horizon 2020. Πρέπει λοιπόν καλύτερα ένα δις να πάει εδώ και τα υπόλοιπα να πάνε στον, τα δύο στον προϋπολογισμό Horizon 2020 για να χρηματοδοτήσουμε προτεραιότητες ε, στα πλαίσια πρόσθετων στόχων που έχω βάλει που είναι ε, θα πρέπει να βάλουμε στην έρευνα πάλι το θέμα της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης που υπήρχε σε προηγούμενα προγράμματα αλλά ειδικά δεν αναφέρεται εδώ στην πρόταση της Κομισιόν και επίσης είναι σημαντικό για την Επιτροπή μας να συμπεριληφθεί. Έτσι λοιπόν έχω μια ειδική μνήμα στην πολιτιστική κληρονομιά στον κανονισμό. Δεύτερον, ως αποτέλεσμα των νέων αρμοδιοτήτων στον αθλητισμό θέλω να αναδείξω τη δυναμική της έρευνας στον αθλητισμό ως μέσον για να βελτιωθεί γενικά η υγεία των πολιτών της Ευρώπης. Επίσης η κοινωνική συνοχή και η ένταξη ε, ενισχύονται. Επίσης τίνεται ο ρόλος των γυναικών στην επιστήμη και την τεχνολογία και ο ρόλος της ακαδημαϊκής έρευνας ε, για, την, για τα νέα προϊόντα και νέα επιχειρηματικά μοντέλα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εκτό, επίσης, σε πρόσβαση στη χρηματοδότηση πρέπει να είναι η πρόσβαση απλούστερη, ευκολότερη και το Horizon 2020 θα πρέπει να μορφούται με το στόχο του Εράσμους θα ήθελα να ακούσω και τις γνώμες των σκιωδών και των άλλων συναδέλφων στην Επιτροπή, που επίσης μου κοινοποίησαν τις απόψεις τους και βοήθησαν πολύ να καταρτιστεί η τωρινή έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Μπάγκο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μακλάρκιν για την γνωμοδότησή της. Έχουμε συζητήσει διάφορα θέματα και με τη βοήθεια της γραμματείας. Θα ήθελα να ξαναδεί το θέμα της ε, μείωσης του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Συντήτου Έρευνας. Γιατί η αφαίρεση 2 εκατομμυρίων από τον προϋπολογισμό θα καταστήσει ανέφικτη τη λειτουργία. Έχουμε... Ε, ένα ποσό που δεν θα πρέπει να αφαιρεθεί από τον προπολογισμό του Τεχνολογικού Ινστιτούτου. Παρακαλώ να το ξανασκεφτεί η συγκεκριά. Ο κύριος Τάκουλα. Ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ σύντομος. Πολύ λίγα σχόλια έχω γιατί δεν βλέπω πώς θα μπορούσα να συμβάλλω στη συζήτηση παρά μόνο ποσοτικά. Είμαι πλήρως ικανοποιημένος από τις αδρές γραμμές της πρότασης της κυρίας Μακλάρκιν και της ιεράρχηση των προτεραιοτήτων προκειμένου να επικεντρωθούν οι πόροι σε ορισμένους τομείς. Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα αυτή η έμφαση που δίνεται στον αθλητισμό. Γιατί πιστεύω και εγώ ότι ο αθλητισμός είναι ένας τομέας πολιτικής που εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Επιτροπής μας και ένας τρόπος να βελτιώσουμε μέσω της προαγωγής του αθλητισμού τη δημόσια υγεία. Άλλωστε, ο αθλητισμός έχει και κοινωνικό ρόλο που δεν θα πρέπει να τον ξεχνούμε. Το ίδιο ισχύει και για την ισότητα των ευκαιριών. Γιατί δυστυχώς ε, στον τομέα αυτό πολλές χώρες υστερούν. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις περικοπές στον προϋπολογισμό συμφωνώ για τον προβληματισμό προς το Τεχνολογικό Ινστιτούτο, γιατί το Τεχνολογικό Ινστιτούτο είναι περισσότερο δίκτυο παρά Προτιμούμε ένα τέτοιο χαλαρό δίκτυο, γιατί τα τεχνολογικά Ινστιτούτα και τα πανεπιστήμια ήδη υπάρχουν. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι μια καλή δικτύωση μεταξύ τους. Επαναλαμβάνω, γενικώ είμαι πολύ ικανοποιημένο από την γνωμοδότηση. Θα καταθέσω καμιά δύο τροπολογίε. Πάντω πιστεύω ότι ήταν πολύ αξιόλογο το έργο της ηγετριάς μας, κυρίας Μακλάρκιν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και εγώ υπογραμμίζω αυτό που είπε ο κύριος Στάκουλα για τον αθλητισμό και εγώ θέλω τους παράγοντες ε, του τρόπου ζωής, lifestyle factors, το ποτό, το τσιγάρο, τα hamburgers, και τα συνεχή fast food. Αυτά όλα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Αλλά ακούγονται στα γερμανικά παράδοξα, αν μεταφράσουμε το lifestyle. Το lifestyle ακούγεται πολύ ωραία στα αγγλικά, όχι όμως στα γερμανικά. Το lifestyle έχει μια θετική έννοια στα αγγλικά, ενώ εδώ εννοούμε κάτι αρνητικό. Οπότε θα πρέπει ίσως να το περιγράψουμε διαφορετικά. Ίσως στα αγγλικά να συνηθίζεται αλλά στα γερμανικά δεν ακούγεται καλά. Α είναι, συμφωνώ και με τον συνάδελφο Μπάγκο, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο έχει αρχίσει τις εργασίες του. Η εργασία του απεδείχθη εξαιρετική και τώρα διευρύνεται και στοχεύει περισσότερο στις δραστηριότητες και οι ΜΜΕ παίζουν ρόλο εδώ. Έτσι λοιπόν η περικοπή που προτείνεται εδώ, δηλαδή από τρία εκατομμύρια σε ένα εκατομμύριο, ε, δεν νομίζω ότι μπορεί να το ισχυριστεί κανείς, θα καταρρεύσει το Ινστιτούτο. Οι διαβουλεύσεις έδειξαν ότι ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες και απαιτήσεις στο Ινστιτούτο αυτό ότι μετά την ε, δρομολόγησή του εργάστηκε πολύ καλά, γι' αυτό δεν πρέπει να είμαστε τόσο αυστηροί εδώ απέναντί του όπως προτείνει η ΕΜΑ. Θα υπάρξει κάποια τροπολογία, να γίνει ίσως μία περικοπή, αλλά όχι αυτού του εύρους. Αυτή ήταν μια σύντομη παρατήρηση από μένα. Δεν είμαι συνεισηγήτρια ούτε σκιώδης βέβαια. Κατά τα άλλα, Συμφωνώ με τις προτάσεις της κυρίας Μακλάρκιν. Υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις. Α, η Κομισιόν. Παρακαλώ, Κομισιόν. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να κάνω κάποια σχόλια. Η ε, η συγκήτρια μίλησε για τη σημασία της αριστείας και της επιστήμης, που είναι και η ακρογωνία η λύθη της πρότασης αυτής, γιατί έτσι θα ενισχύσουμε την ιδέα ότι το πρόγραμμα πλαίσιο θέλει να στηρίξει τις καλύτερες ερευνητικές ομάδες και την, να προωθήσει την αριστεία στην Ευρώπη. Προτάθηκαν αυξήσεις στο προπολογισμό. Είπατε ότι είστε υπέρ του προπολογισμού και μάλιστα ζητάτε και αύξηση, παρά είναι φιλόδοξα νομίζω τα σχόλιά σα. Τώρα για τα υπόλοιπα σημεία αναφέρθηκα προηγουμένω στο γεγονός ότι η πολιτιστική κληρονομιά ήδη καλύπτεται από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συνεχίζεται πολύ διεξοδική συζήτηση για το θέμα αυτό και στο Συμβούλιο. Επίσης αναφέρθηκαν τα θέματα του τρόπου ζωής, του lifestyle, ε, από ευκαιρία του αθλητισμού. Οι δημογραφικές αλλαγές, η υγεία και το θέμα της ευημερίας περιλαμβάνονται στην πρόταση, τουλάχιστον μερικές πτυχές. μπορούμε να τις συνδέσουμε με τον αθλητισμό. Είναι πολύ σε αυτή η διασύνδεση αθλητισμού και τρόπου ζωή, υγεία κτλ. Επίσης προτείνεται μείωση του προπολογισμού του Τεχνολογικού Ινστιτούτου δεν ε, κατάληξαμε ελαφρά την καρδία στο ποσό αυτό. Ήταν πολύ διεξοδική η πρόταση και πολύ χρονοβόρα η διαδικασία της επεξεργασίας της με εκτενείς διαβουλεύσεις και υπήρξε υποστήριξη της πρότασης. Γνωρίζω ότι ο συνάδελφος, της Γενικής Διεύθυνσης για, για τον πολιτισμό και την παιδεία θα ήθελε να πει δύο λόγια ειδικά για το θέμα αυτό, αν δεν έχετε αντίρρηση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ ε, για την γνωμοδότηση που έχετε καταθέσει. Το Τεχνολογικό Ινστιτούτο στηρίζεται σε υπάρχουσα αριστεία και το γεγονός ότι έχει συμπεριληφθεί στον ορίζοντα 2020 ακριβώς ε, οφείλεται στη δυνατότητα συμπληρωματικότητας και συνέργειας που έχει να αντιμετωπίσει αυτές τις ε, προκλήσεις της κοινωνίας. Γιατί ε, η, ακριβώς η κοινωνία της γνώσης προωθείται μέσω της ικανοποίησης των κοινωνιακών προκλήσεων στις οποίες συμβάλλει και το Τεχνολογικό Ινστιτούτο. Είπατε ότι δεν θα επιτύχει τη μόχλευση το Τεχνολογικό Ινστιτούτο και ότι δεν θα, δεν θα μπορέσει να συγκεντρώσει την κρίσιμη μάζα για να, να υλοποιήσει τους στόχους του αν μειωθεί ο προπολογισμό. Όλοι γνωρίζουμε ότι το Τεχνολογικό Ινστιτούτο δεν α, λειτουργήσε για πολύ καιρό. Πάντως μετά την αξιολόγηση που έγινε είναι θετικά τα πρώτα αποτελέσματα. Γι' αυτό ακριβώς και καταλήξαμε σε πολύ αυστηρέ προϋποθέσεις προκειμένου να απελευθερωθεί ο προπολογισμό και μάλιστα σε δύο δόσεις. Αρχικά την πρώτη και έπεται και δεύτερη δόση του προϋπολογισμού που θα εκταμιευθεί μόνο μετά από θετική έκβαση, θετική αξιολόγηση της ενδιάμεσης ε, αναθεώρησης. Θέλουμε ακριβώς να συνεχίσει τη ορθή πορεία το Τεχνολογικό Ινστιτούτο και από αυτό εξαρτάται η εκταμίευση της δεύτερης δόσης. Νομίζω ότι πολύ καλό μέτρο αυτό, οι δύο δόσεις, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των δράσεων του Τεχνολογικού Ινστιτούτου, όπως είπατε και εσείς. Ναι, νομίζω ότι είναι και στο διατακτικό. Δεν είναι μόνο δηλαδή αυτό μια φιλική κουβέντα. Ωραία, ο κύριος Μπόρις. Ε, Ευχαριστώ. Ε, το τεχνολογικό Ινστιτούτο, αν θέλουμε να είναι αποτελεσματικό στην καινοτόμο δράση του και αν θέλουμε να γίνει μοχλός ε, και ατμομηχανή για καινοτόμα σχέδια στον ορίζοντα 2020, που είναι πολύ φιλόδοξα και γνωρίζουμε πόσο φιλόδοξη είναι η στόχη της στρατηγική 2020, δεν μπορεί να στερήσουμε ε, το Ινστιτούτο από τον προπολογισμό. Θα διαφωνήσω λοιπόν με τους συναδέλφους. Έγιναν πολλές προσπάθειες για να λάβουμε εμεί την έδρα, τελικά ανατέθηκε στην Ουγγαρία. Ε, είναι πολύ σημαντικό αυτό το δίκτυο και θα εξασφαλίσει συνεργασία στην Ευρώπη και με ένα επαρκή προπολογισμό θα μπορέσει να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση πόλος ενδιαφέρον και ονοτόμων προγραμμάτων. Είμαι υπέρ λοιπόν του προπολογισμού και κατά της μείωσης. Ό,τι αφορά τις ε, ερωτήσεις ε, της Επιτροπής Αθλητισμού και Παιδείας. Για πρώτη φορά κάποιο πρόγραμμα του ορίζοντα 2020 θα περιλάβουν και κάποιες ανθρωπιστικές επιστήμες και κάποιους κοινωνικούς στόχους. Αυτή είναι μια καινοτομία του ορίζοντα, γιατί στο παρελθόν δεν προβλεπόταν τέτοια σχέδια. Τώρα, χάρη στο νέο κανονισμό, θα μπορέσουμε να, να ε, επενδύσουμε και στις κοινωνικές επιστήμες και στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Αυτό είναι μια καινοτομία στην ιστορία, κοινωνικές επιστήμες, στην επιστήμη, πέραν του αθλητισμού, περιλαμβάνονται και αυτά τα θέματα. Δυστυχώς στην πρόταση του Συμβουλίου δεν υπάρχουν διεξοδικές προτάσεις. Αναφέρεται μόνο αυτό το σύνθημα, ανθρωπιστικές επιστήμες, κοινωνικές επιστήμες, αλλά τίποτα συγκεκριμένο. Μπορούμε λοιπόν να υποστηρίξουμε και σε αυτό το σημαντικό τμήμα των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών μέσω της καινοτομίας και της τεχνολογίας ή τουλάχιστον με κάποιο άλλο τρόπο με κάποιες άλλες δραστηριότητες ε, για τις κοινωνικές δράσεις. Θα μπορούσατε να δώσετε μία απάντηση ως προς αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω. Η Κομισιόν έχει να απαντήσει, μπορεί να απαντήσει στην ερώτηση αυτή. Η εκπρόσωποι της Κομισιόν. Uh, Σκεφτούμε παρακαλώ, μπορούμε και θα σας απαντήσουμε. Έχετε χρόνο. Κυρία Μακλάρκιν, παρακαλώ, στο κείμενό σας προσέξτε την τροπολογία 6 για να, να μην γράφει να συμμορφούνται με το πρόγραμμα Εράσμους, αλλά γενικότερα με τα προγράμματα εκπαίδευσης. Μην αναφερθούμε συγκεκριμένα στο όνομα, γιατί υποθέτουμε ότι δεν θα είναι και το σωστό. Μπορεί να μην συμφωνείτε, αλλά εγώ το πιστεύω. Είτε λοιπόν εσείς θα επανέλθετε μόνοι σας και θα μιλήσετε για προγράμματα εκπαίδευσης ή θα ε, παρέμβω εγώ με τροπολογία. Και πότε θα μας απαντήσει η Κομισιόν. Πότε θα απαντήσετε στην ερώτηση του κυρίου Μπόρις. Γραπτός, εγγράφος θα απαντήσετε. Πώς θα απαντήσετε. Εντάξει, εγγράφος. Θα λάβουμε γραπτός την απάντηση. Έμα. Ευχαριστώ. Σημείωσα τα σχόλιά σας. Όλοι οι συνάδελφοι έκαναν καλά σχόλια, τους ευχαριστώ. Για αυτό του... που είπε ο Ούγκρος συνάδελφος για το Τεχνολογικό Ινστιτούτο. Ο προϋπολογισμός του Ινστιτούτου είναι 309 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή. Η προτινόμενη αύξηση είναι στα 3 δις. Ε, η πρότασή μου να φτάσει στο 1 δισεκατομμύριο ούτως ή άλλως αποτελεί τεράστια αύξηση χρηματοδότησης του Ινστιτούτου. Ε, όπως ακούσαμε ή δεν ακούσαμε <laughs> σήμερα. Είναι ένα καινούριο ίδρυμα και δεν ξέρουμε πόσο αποτελεσματικό θα είναι. Ε, πώς θα χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά αυτά τα τρία δις που είναι πάρα πολλά. Θέλουμε λοιπόν Δείτε λοιπόν την τροπολογία μου που ούτως ή άλλως η χρηματοδότηση αποτελεί τεράστια, προβλέπει τεράστια αύξηση. Δηλαδή από τα 309 εκατομμύρια φτάνουμε στο 1 δις. Σας ευχαριστώ για τα όσα είπατε για τον αθλητισμό. Ευχαριστώ Πρόεδρε για το σχόλιο σας, το σχόλιο σας και τον τρόπο ζωής. Ε, προσπαθώ να τα εντάξω όλα αυτά στους πυλώνες που υπάρχουν ε, στον προϋπολογισμό του ορίζοντα. Ε, προκλήσεις στην, ε, που αντιμετωπίζει η κοινωνία. Μία από τις προκλήσεις είναι ακριβώς αυτή. Προσπαθούμε να το εντάξουμε λοιπόν. Εμείς προσπαθούμε η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή ε, να λάβει υπόψη τα δικά μας σχόλια. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι όταν θέλουμε να προωθήσουμε κάποια πράγματα. Και ευχαριστώ για την Κομισιόν που μας είπε ότι αυτή τη στιγμή συνεχίζεται η συζήτηση σε ό,τι αφορά την πολιτιστική κληρονομιά και φαντάζομαι ότι θα συμφωνείτε ότι πρέπει να γίνει μια συγκεκριμένη αναφορά σε ό,τι αφορά αυτή την πολιτιστική κληρονομιά. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι πολεμούμε πάρα πολύ συγκεκριμένα και στοχευμένα ε, για το θέμα του οικονομικού. Το, θέμα το, οικονομικό. Και το, που, και το θέμα του πού βρίσκουμε τα κονδύλια. Ωραία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπάγκο ζητεί πάλι το λόγο. Δεν έχουμε πάρα πολλά θέματα σήμερα που λείπουν τόσο πολύ, οπότε μπορεί να ξαναμιλήσει ο κύριος Μπάγκο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για τη γενεοδορία σας, μία πρόταση θέλω να προσθέσω. Είναι ένα παιχνίδι με τα νούμερα αυτό τελικά. Το θέμα όμως πέρα από τα νούμερα ε, υπάρχουν και λεπτομερή προγράμματα. Οι εμπειρογνώμονες έκαναν υπολογισμούς για αυτό το ποσό. Δεν νομίζω ότι πρέπει εδώ να, συνεχί... αρχίσουμε μια πολιτική συζήτηση. Θέλω να καταφέρουμε να φτάσουμε σε συμβασμό ως προς το θέμα αυτό των... του ποσού. Θα γίνει αυτό στην πορεία της συζήτησης, είναι άλλωστε πολύ προσεκτική και η Κομισιόν λέει θα πληρώσει σε δύο δόσεις. Δεν είναι τόσο βέβαιη και εκείνη ότι θα ε, απορροφηθούν αυτά που έχει προβλέψει. Οπότε πράγματι γιατί να είναι τόσα πολλά τα χρήματα αν και η ίδια δεν πιστεύει στην απορρόφηση. Θα το ξαναδούμε αυτό. Νομίζω όμω ότι η συζήτηση σήμερα έθιξε το θέμα αυτό τουλάχιστον και σε συμφωνία μεταξύ όλων μπορούμε να βρούμε μια συμβιβαστική λύση με την κυρία Μακλάρκιν και με του άλλου συναδέλφου και τι άλλε πολιτικέ ομάδε. Λοιπόν, τελειώνει η συζήτηση. Σε αυτό το σημείο έχουμε μια προθεσμία 7 Ιουνίου για την κατάθεση τροπολογιών. Έμα, το χρονοδιάγραμμα ήθελα να πω. Ελπίζουμε να έχουμε ακόμα μια συνάντηση των σκιωδών εισηγητών. Στις 7 Ιουνίου για τις τροπολογίες θα ψηφίσουμε και θα ψηφίσει η αρμόδια επιτροπή στις, το πρωί στις 10 Ιουλίου. Κοντεύει η 7η Ιουνίου, την επόμενη εβδομάδα είναι. Οπότε να βιαστούμε να καταθέσουμε τις σημαντικότερες τουλάχιστον τροπολογίες. Εντάξει λοιπόν, 12 το μεσημέρι, 7 Ιουνίου. Κλείνει η συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ την ΕΜΑ και περνάμε στο σημείο 5, τροποποίηση της οδηγίας για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα. Θεέ μου. Η Ζαμπίνε Φερχάιεν, έχει το λόγο. Όχι, δεν είναι και τόσο τρομερά τα πράγματα. Πρόκειται για την τροπολογία οδηγίας από το 2003 που ρυθμίζει πώς ε, θα χρησιμοποιηθεί η ε, πρόταση. Καταρχήν ε, η κοινή γνώμη έχει δικαίωμα ε, σε πληροφορίες που θεωρούνται και από την Κομισιόν δημόσιο αγαθό και θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση στην κοινή γνώμη αλλά και να διατίθενται για περαιτέρω εμπορική χρήση. Εδώ η Κομισιόν βλέπει ένα τεράστιο δυναμικό κοινωνικό και εις ό,τι αφορά τις ε, καινοτομίες και εις ό,τι αφορά το γλάβε του πολιτισμού νομίζω ότι πολλά έχουμε να αποκομίσουμε. Εγώ είμαι υπέρ των βημάτων προς, την, προς το μόνιμο άνοιγμα και την διαρκή πρόσβαση στις πληροφορίες και την ψηφιοποίηση των ε, πολιτιστικών δεδομένων που διευκολύνει ακόμη περισσότερο την πρόσβαση και σε βιβλιοθήκες πανεπιστημιακές και όχι σε μουσεία, νομίζω ότι είναι μια καλή προσέγγιση. Η πρόταση οδηγίας όμως έχει ορισμένα θέματα που χρειάζονται διευκρινήσεις θεωρώ και δεν ε, είναι τόσο ξεκάθαρα τα θέματα από ό,τι έδειξαν και οι συζητήσεις με την Κομισιόν. Αυτά θα πρέπει να τα δούμε στο κείμενο, διότι αν δεν γίνουν διευκρινήσεις θα υπάρξουν επιπτώσεις δημοσιονομικές στους δημόσιους φορείς και θα υπάρξουν και αρνητικές επιπτώσεις στην προσπάθεια ψηφιοποίησης στον πολιτιστικό τομέα περιοριστικά μέτρα αναχρηματοδότησης που πρότεινε η Κομισιόν. Στη γνωμοδότησή μου λοιπόν έχω θέσει πέντε ε, προτεραιότητες. Καταρχήν ότι η εξουσία λήψης αποφάσεων σχετικά με το ποια θα είναι τα κοινοποιούμενα δεδομένα ε, θα είναι των δημοσίων ε, φορέων ε, που θα αποφασίζουν για την δημοσιοποίηση των δεδομένων. Θα πρέπει δηλαδή οι εθνικές αρχές να έχουν την εξουσία αυτή. Επίσης ορισμένα έγγραφα μπορεί να αποκλείονται από την περαιτέρω χρήση τους γιατί πολλά πρώτα δεδομένα δεν έχουν ε, τύχη επεξεργασίας ούτε έχουν υποστεί έλεγχο. Θα πρέπει να ε, υπάρχει μια επεξεργασία δεδομένων περαιτέρω και όταν δημοσιεύονται όλα τα δεδομένα ε, στα πλαίσια της ε, οδηγίας προστασίας δεδομένων δημιουργούνται κάποιοι κίνδυνοι. Ένα δεύτερο θέμα είναι η διαλειτουργικότητα. Εδώ πρέπει να υπάρξουν σαφείς διατυπώσεις, να είναι ξεκάθαρο ότι οι δημόσιες αρχές δεν υποχρεούνται να παρουσιάζουν ε, σε ψηφιακή μορφή όλα τα μεταδεδομένα γιατί διατίθενται ε, αφενός ε, διότι συμφωνούμε με την Επιτροπή ότι μόνο τα δεδομένα που διατίθενται ήδη σε ψηφιακή μορφή θα έπρεπε να διατίθενται σε τεχνολογικά ουδέτερες μηχαναγνώσιμες μορφές. Ε, αλλιώς θα υπάρξουν ε, οικονομικές υποχρεώσεις που κανείς δεν θα μπορέσει να υπομιστεί, Πόσο μάλλον που δεν θα υπάρχει και ξεκάθαρο όφελος από όλο αυτό. Σημαντικό είναι και η τεχνολογική ουδετερότητα, όπως είπαμε, να, μην, να είναι σαφές δηλαδή ε, ότι θα πρέπει να είναι δεδομένα προς βάσιμα σε όλους. Επίσης η σύσταση ανεξάρτητη της αρχής, ε, ε, αυτό είναι ένα αίτημα ε, πολύ σημαντικό. Ε, θα πρέπει να προσέξουμε να μην είναι όλα αυτά αντίθετα προς τις προσπάθειες των κρατών μελών για μείωση της γραφειοκρατίας, για δημοσιονομική εξυγίανση. Ε, πολλές φορές αναφέρεται και η σύσταση ανεξάρτητων αρχών. Εγώ νομίζω ότι ανάλογα με τη δομή σε κάθε κράτος μέλος ε, μπορούν αντίστοιχα να ε, προβλεφθούν οι καταλληλότερες υπηρεσίες και κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να παρακολουθεί με το δικό του τρόπο πώς θα εφαρμόζεται η οδηγία. Οι δημόσιες διοικήσεις Ε, θα έχουν να υπομισθούν ε, μεγάλο φόρτο εργασίας όταν πρόκειται για το βάρος της απόδειξης, ε, όταν υπάρχουν προβλήματα και επίμαχες υποθέσεις θα πρέπει να, να αποδεικνύεται αν για παράδειγμα η... το μουσείο ή η βιβλιοθήκη, πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη ετήρησε όλες τις διατάξεις και έχει ε, κοινοποιήσει όλα τα έγγραφα και ε, πάντοτε θα πρέπει να υπάρχει η απόδειξη ότι όλα έχουν γίνει σωστά. Αν υπάρχει κριτική θα πρέπει να αιτιολογείται αυτή και όχι να ε, υποχρεώνει τις αρχές αυτές να ε, επομίζονται το βάρος της απόδειξης. Το τέταρτο θέμα ε, είναι τα τέλη και οι αρχές χρέωσης. Εδώ ε, για την εμπορική περαιτέρω χρήση των δεδομένων οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να, επιβάλλουν, να μπορούν να επιβάλλουν ανταποδοτικά τέλη και αρχές χρέωσης για την ποιότητα της πληροφόρησης του δημόσιου τομέα και για Πολύ συχνά η ψηφιακή μορφή συνδέεται με υψηλά κόστη και τα κόστη αυτά θα πρέπει όταν πρόκειται και για εμπορική χρήση θα πρέπει να καλύπτονται από τα τέλη και τις, αρχές, τις χρεώσεις. Επίσης τα αρχεία των βιβλιοθηκών εν μέρη χρηματοδοτούνται από τις ίδιες τις ε, βιβλιοθήκες και πολλές φορές δημιουργούνται ελλείμματα τα οποία δεν ε, ε, είναι μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε τοπικό επίπεδο. Ε, οι δήμοι, οι κοινότητες, πολλές φορές δημιουργούν ελλείμματα. Εδώ θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα αναχρηματοδότησης. Το πέμπτο σημείο είναι οι συμφωνίες αποκλειστικότητας, ιδιαίτερα στον τομέα του πολιτισμού. Έχουν μεγάλη σημασία. Ε, έχουμε εδώ αναφερθεί σε διάφορες πρωτοβουλίες ψηφιοποίησης. Πολλές φορές έχουμε ιδιωτικέ συμπράξεις και ένας ιδιώτης εταίρος μπορεί να αναλάβει την ψηφιοποίηση και έχει το δικαίωμα αποκλειστικά για ένα χρονικό διάστημα να μπορεί να εμπορεύεται το αποτέλεσμα αυτό. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να επιτρέπεται αυτό, είναι προς το συμφέρον της κοινή γνώμης, γιατί έτσι μπορεί να επιταχυνθεί πάρα πολύ η διαδικασία της ψηφιοποίησης. Όμως θα έλεγα ότι σε αυτή την περίπτωση η συμφωνία αποκλειστικότητας θα πρέπει να περιορίζεται σε 7 χρόνια. Είναι ένας ε, συντελεστής αναχρηματοδότησης, ε, ο οποίος ε, είναι πολύ λογικός και μετά από 7 χρόνια θα πρέπει να είναι δημόσια η υπηρεσία αυτή. Έτσι μπορούμε με ε, έξυπνο τρόπο να επιταχύνουμε και να προωθήσουμε τη διαδικασία της ψηφιοποίησης. Η έκθεση όπως είδα από χθε ή από σήμερα ε, έχει μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες που χρειαζόμαστε γιατί ήταν λίγο δύσκολο αυτό να γίνει, ε, επειδή είχαμε και τη χθεσινή γιορτή. 7 Ιουνίου είναι η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών. Ε, θα ήθελα να κάνουμε στις 4 Ιουνίου το βράδυ μια συνεδρίαση των σκιωδών, μια μέρα πριν από τη συνεδρίασή μας, αλλά θα πρέπει να συνεννοηθώ με τους σκιώδεις, ίσως θα πρέπει να αλλάξουμε την προθεσμία. 10 Ιουλίου θα είναι η συνεδρίαση της Επιτροπής και η Ήτρε που είναι αρμόδια επί της ουσίας θα ψηφίσει στις 24 Σεπτεμβρίου. Ευχαριστώ. Είναι πολύ σύνθετο το θέμα αυτό και έχει πολύ χαίρομαι που δεν χρειάζεται να τον αλάβω εγώ και να ασχοληθώ. Ευχαριστώ τη Ζαμπίνη που ασχολήθηκε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ Ζαμπίνη που έκανε όλον αυτόν τον κόπο. Δεν έχω να προσθέσω πολλά σε αυτά που είπες. Ε, θεωρώ ότι καταρχήν είναι σωστό αυτό που λες, ότι ε, δεν ε, θέλουμε να δημιουργήσουμε μια μεγάλη υπηρεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να ασχοληθεί με το θέμα, αφήνουμε τα κράτη-μέλη να βρουν σωστές λύσεις, αφού άλλωστε υπάρχουν ε, ήδη δομές στα κράτη-μέλη που μπορούν να, λάβουν τα θέματα αυτά. Και εν πάση περιπτώσει υπάρχουν ε, στη διάθεσή μας και νομικά μέσα επίλυσης του θέματος σημαντικό είναι ότι αναφέρεται αυτό ότι δεν θα εφαρμόζεται στη δημόσια ραδιο, στην κρατική ραδιοφωνία η οδηγία αυτή. Αυτό είναι σημαντικό γιατί ε, είναι διαφορετικά διαφορετικός ο τομέας αυτός και δεν νομίζω ότι θα πρέπει να καλύπτεται από αυτή την οδηγία. Επίσης ε, για τα τέλη και τις αρχές ε, χρέωσης και εδώ είναι αναγκαίο να προβλεφθεί αυτό για όλους τους δημόσιους φορείς και εν ώψη των οικονομικών τους. Ε, είναι σημαντικό να τονίσουμε τον ανταποδοτικό χαρακτήρα αυτών των τελών και ε, στην οδηγία θα πρέπει να αναφέρεται ξεκάθαρα τι επιτρέπεται αλλά και τι όχι. Σε ό,τι αφορά τις συμφωνίες αποκλειστικότητας θα πρέπει να το σκεφτώ λιγάκι αν έτσι όπως το παρουσίασε στο θέμα με βρίσκει σύμφωνη, αλλά ε, θα δω τη μετάφραση αύριο και θα μπορέσω να δω όλες τις λεπτομέρειες. Αλλά ακούγοντα αυτά που μας είπες, νομίζω ότι έχουμε μια καλή βάση για την περαιτέρω συζήτηση και θεωρώ ότι θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία που θα οδηγήσει σε μια ωραία ε, γνωμοδότηση και θα τη δώσουμε στην Επιτροπή Ήτρε. Ευχαριστώ. Ζαμπίνε, πού είναι αυτή η υπηρεσία μαμούθου δεν τη θέλεις, γιατί εγώ δεν τη βλέπω, αναφέρεται γενικά ότι θα πρέπει και σε επίπεδο νοσιακό να διασφαλίσουμε την επιτυχία του εγχειρήματος, θα πρέπει να υπάρξει συντονισμός των εθνικών αρχών. Δεν λέει τίποτα για μια υπηρεσία μαμούθ. Βέβαια, ε, φαντάζομαι ότι κάπου θα είναι, δεν το βρήκα γιατί υπάρχουν πολλές υπηρεσίες έτσι κι αλλιώς και συμφωνώ ότι δεν χρειάζεται, αλλά στο σημείο 14 δεν το βλέπω ή μήπως δεν διαβάζω καλά. Σαμπίνε. Η υπηρεσία Μαμούφ δεν αναφέρεται ως έτσι κυριολεκτικά, αλλά αναφέρεται ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί μια αντίστοιχη αρχή. Και θα ήθελα διευκρίνηση να μας πούν ότι δεν θα δημιουργήσουν νέα υπηρεσία, αλλά οι φυστάμενοι φορείς θα αξιοποιηθούν. Πού δηλαδή είναι αυτό. Στο 14 του το τροποποίησης δεν αναφέρεται για μια νομότυπη εφαρμογή κάποιες διατάξεις αυτής της οδηγίας κλπ. κλπ. Η εποπτεία θα πρέπει να υπάρχει από ανεξάρτητες αρχές. Αρχές, όχι αρχή. Ε, θα χρειαστεί συντονισμός επίσης αυτών των ανεξάρτητων αρχών. Πληθυντικός αναφέρεται. Δεν υπάρχει αυτή η απειλητική υπηρεσία μαμούθα. Δεν θα είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο μία, δηλαδή δεν θα πρέπει να είναι κεντρική αρχή. Εγώ απλώς ζήτησα μια διευκρίνηση εδώ, ότι μπορούν και οι φυστάμενες αρχές να το αναλάβουν και ότι θα πρέπει τα κράτη-μέλη τα ίδια να αποφασίζουν πώς θα το χειριστούν, γιατί υπάρχουν ε, τέτοιες, ε, τέτοιοι φορείς. Να θέλω αυτή τη διευκρίνηση, ότι δεν θα δημιουργηθεί χωριστή καινούργια αρχή. Είπα ότι έκανα πολλές συζητήσεις με την Κομισιόν. Πρόκειται για διευκρινήσεις, ούτως ώστε να είναι ξεκάθαρες οι δηλώσεις των Κομισιόν και να μην θεωρήσουν τα κράτη-μέλη ότι θα πρέπει τώρα να δημιουργήσουν καινούριε αρχές. Δηλαδή προληπτικά δράσε για να προλάβεις κάτι που μπορεί να έχει στο μυαλό του κάποιος. Αλλά η Κομισιόν μπορεί να μην το έχει υπόψη της αυτό να το κάνει. Πάντως θετικό είναι ότι το ε, αναφέρει αυτό προληπτικά. Η Κομισιόν ε, εκπροσωπείται. Ο κύριος Ρίτσαρτ Σουίτενχαμ. Πρισνιεύσκα. Όχι. Καλώς, τι να κάνουμε, τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε. Α, θα προχωρήσουμε χωρίς ε, ε, σας. Μας λείψατε σήμερα. Α, η κυρία Βενέρα Πατού. Ένα ερώτημα. Ποιο είναι το πεδίο εφαρμογής αυτού του ψηφίσματος. Αφορά και τα δημόσια δεδομένα και τα, και τα ιδιωτικά στοιχεία των πολιτών. Äh, η, οδηγία δεν λέει τίποτε για το ποια θα είναι τα δημοσιευόμενα δεδομένα. Αναφέρει τη μορφή που θα έχουν αυτά τα ε, δεδομένα που θα κοινοποιούνται και είναι διαφορετική και συνδυασμένη η νομοθεσία στα κράτη-μέλη από το 2003 ή στηρίζεται στην εφαρμογή της οδηγίας για να κριθεί η ποιότητα των δεδομένων που θα κοινοποιούνται. Ε, εδώ αναφέρονται τα προσωπικά δεδομένα που αποκλείονται, ε, ισχύουν οι κανόνες προστασίας δεδομένων, δεν μπορούν να ε, δημοσιεύονται όλες οι λεπτομέρειες προσωπικών δεδομένων κάθε πολίτη. Τα δεδομένα που θα δημοσιεύονται θα ψηφιοποιούνται ε, για να μπορούν να ε, εξυπηρετούν κι άλλες χρήσεις εμπορικές για την περαιτέρω ε, ανάπτυξη καινούριων υπηρεσιών όταν έχουμε ας πούμε δεδομένα κτηματολογίου μπορώ να τα διαθέσω σε γεωφυσικές υπηρεσίες μέσα από εφαρμογές ή να τα αξιοποιήσω με καινούργιες εφαρμογές. Έτσι δημιουργείται προστιθέμενη αξία και η Κομισιόν υπολογίζει σε κάποια δισεκατομμύρια ε, προστιθέμενης αξίας με τις νέες εφαρμογές και τις νέες υπηρεσίες που θα δημιουργηθούν έτσι. Δεν πρόκειται όμως για προσωπικά δεδομένα που τα προστατεύει η νομοθεσία προστασίας δεδομένων. Ναι, ναι, ναι, δεν θίγονται αυτά. Πρόκειται για την νέα χρήση ε, δεδομένων που μπορεί να τύχουν περαιτέρω εφαρμογής. Δεν ζητεί άλλο τον λόγο, οπότε τελειώνουμε και το... Α, 11 Ιουνίου προθεσμία κατάθεση τροπολογιών, το μεσημέρι. 11 Ιουνίου το μεσημέρι. Και τον Ιούλιο θα γίνει ψηφοφορία. Ωραία. Προχωρούμε. Επόμενη έκθεση της ΕΜΑΣ, έκθεση σχετικά με την εφαρμογή αποτελέσματα της οδηγίας για το δικαίωμα παρακολούθησης. ΕΜΑ, παρακαλώ. Ευχαριστώ ξανά, Πρόεδρε. Αυτή η έκθεση αφορά την ε, εισαγωγή του δικαίωματος παρακολούθησης και την ε, επίπτωση στην ευρωπαϊκή αγορά. Η Επιτροπή μας θα συμφωνήσει ότι η οδηγία ήταν επιτυχία και επιτρέπει στους ε, καλλιτέχνες να παρακολουθούν, να παρακολουθούν την, την πορεία των έργων τους και αναγνωρίζει την αξία των πολιστικών αγαθών. Ε, το θέμα είναι όμως ε, ότι μειώθηκε πάρα πολύ ε, το μερίδιο της αγοράς ε, παγκόσμια της Ευρώπης γιατί υπάρχει ένα τεράστιο διοικητικό άχθος στους ε, πολίτες και υπάρχει εμπορικό μειονέκτημα σε σχέση με τις τρίτες χώρες. το βάρος είναι ειδικά μεγάλο για τους, για τους μικρούς οίκους δημοπρασίας. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν η Κομισιόν να είναι πιο δραστήρια και να ενθαρρύνει τις τρίτες χώρες να εισαγάγουν το δικαίωμα παρακολούθησης μεταπόλησης και φαντάζομαι ότι δεν έχει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή, δεν έχει αυτή τη δύναμη να επιβάλλει αυτό το δικαίωμα παγκόσμια. Ε, επίσης αυτή την επέκταση του δικαιώματος παρακολούθησης ε, ε, στους μη ζώντες καλλιτέχνες το φοβάμαι. Ειδικά στους μικρούς εμπόρους είναι δύσκολο να βρούμε τους μικρούς εμπόρους και μπορεί το βάρος να είναι πολύ μεγάλο για αυτούς. Θα ήθελα λοιπόν η Κομισιόν να κάνει μία μελέτη αξιολόγηση για την επίπτωση εφαρμογής αυτού του δικαιώματος σε καλλιτέχνες που έχουν πεθάνει. Θέλουμε να έχουμε μια υγιή αγορά εδώ στην Ευρώπη έργων καλλιτεχνικών που θα ε, συνεχίσει αυτόν τον κύκλο δημιουργίας δικαιωμάτων. Και πιστεύω ότι μια τέτοια έκθεση αξιολόγηση θα είναι πολύ σημαντική. Θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις σας ε, για την εκνομοδότηση αυτή τώρα. Δεν βλέπω κανέναν. Θυμάμαι όμως ότι κάποια στιγμή είχα ε, συζητήσει με ανθρώπους που μου παρουσίασαν το θέμα αυτό ότι τα μέτρα αυτά ε, ισχύουν μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι αλλού. Και η αγορά μετατοπίζεται στην Ασία και την Αμερική και χάνουμε πολύ τη θέμενη αξία. Χαίρομαι λοιπόν που ασχολούμεθα τώρα με το ζήτημα αυτό Ελπίζω ότι η ΕΜΑ είναι σε επαφή με την νομική επιτροπή, γιατί ξέρω ότι λένε η πρόεδρος της επιτροπής είχε υποδεχθεί εκείνους τους Εκείνα τα πρόσωπα τα οποία είχαν ε, καταγγείλει την κατάσταση η οποία στραγγαλίζει κυρίως τις μικρές γκαλερί. Ε, θέλω πάρα πολύ λοιπόν να ε, συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση γιατί το, κατα, κατάλαβα τη σημασία του θέματος. Δεν ξέρω, υπάρχουν άλλες γνώμες. Ο Μάρκο. Ο Μάρκος Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για αυτά που μόλις τώρα είπε η κυρία Μακλάρκιν, θα ήθελα να κάνουμε μαζί ένα προβληματισμό. Αυτό το στοιχείο είναι πολύ σημαντικό. Αυτά που ανέφερε είναι πολύ σημαντικά. Και αυτά που είπατε εσείς, Πρόεδρε, για το θέμα της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων. Καλό θα ήταν να δούμε τι άποψη έχουν αυτοί οι συνάδελφοι της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων. Μ' αρέσουν κυρίως αυτά που πρότεινε η κυρία Μακλάρκιν σε ό,τι αφορά την ε, εισαγωγή της έρευνας ε, επί των πολιτιστικών αγαθών στην Ευρώπη. Είναι κάτι που εμείς ως Επιτροπή Πολιτισμού θα πρέπει να το προτάξουμε. Γιατί δεν έχει προβλεφθεί συγκεκριμένα τουλάχιστον στον ορίζοντα 2020. Αυτό το συμμερίζομαι απόλυτα και νομίζω ότι μπορούμε να το, να το ζητήσουμε πιο εμφατικά ακόμα. Ευχαριστώ κύριος Μπάγκο. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με τους προηγούμενους ομιλητές. Είναι ένα ισορροπημένο κείμενο αυτό της ΕΜΑΣ που υπογραμμίζει τα προβλήματα που έχουμε στην ευρωπαϊκή αγορά έργων τέχνης. Η κινέζικη αγορά αυξάνεται. Αυξάνει το μερίδιό της παγκόσμια και η ευρωπαϊκή αγορά μειώνεται. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να δημιουργήσουμε ένα επίπεδο ισότητας. Είναι πολύ σημαντικό να τονίσω στην ε, Επιτροπή ότι πρέπει να εφαρμόσουμε και τους ε, κανόνες στην Ευρώπη. Επίσης, ε, αυτό θα έχει και θετική επίπτωση στην παγκόσμια αγορά. Γιατί θα αναπτυχθούν, θα επηρεάσει ας πούμε και την αύξηση των δεξιοτήτων στην κοινωνία και την απασχόληση εν γέννη. Κοιτάζω προς την κατεύθυνση της Κομισιόν. Τα έδρανα, τα κενά πολλαπλασιάζονται. Κανείς πάλι. Δεν ξέρω, μήπως πρέπει να στείλουμε ένα σημείωμα στην Κομισιόν ότι αποδίδουμε μεγάλη σημασία στην παρουσία τους, έστω και τις μέρες μετά τη γιορτή. Να το αναλάβετε αυτό, γραμματεία. Έμα, Ευχαριστώ για τα σχόλιά σας συνάδελφοι. Και εγώ είμαι απογοητευμένη που δεν είναι εδώ η Επιτροπή για να απαντήσει σε κάποια από τα ερωτήματα που έχουμε, ιδίω για την επίπτωση που έχει αυτό, για την εφαρμογή της, γιατί θέλουμε να έχουμε μια ζωντανή αγορά στην Ευρώπη που δεν θα ε, επηρεάσει ούτε την πολιτιστική μας κληρονομιά, ούτε θα την διώξει το εξωτερικό. Θέλουμε να βρούμε μια λύση στην ε, Ευρώπη εδώ, αλλά να μην στρεβλώνει τα πράγματα, ούτε να μας ε, βγάζει εκτός αγοράς. Θα πρέπει να είναι ισορροπημένη λοιπόν η λύση. Σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. 6 Ιουνίου είναι η ημερομηνία για τις τροπολογίες, μία μέρα νωρίτερα, ε, ούτως ώστε η γραμματεία να μπορέσει να τα συγκεράσει όλα και στις 10 Ιουλίου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τελειώνουμε και το σημείο 6. Το 7 δεν μπορούμε να το καταπιαστούμε γιατί η συγγήτρια ε, ανεξήγητα δεν βρίσκεται εδώ. Κάποιοι άλλοι ε, είπαν ότι... Όχι, έρχεται, έρχεται, έρχεται κυρία Σάκε. Α, τα αποσύρω όλα και χαίρομαι πολύ που θα έρθει. Η ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Θα το συζητήσουμε όταν έρθει το σημείο 8 δεν θα το συζητήσουμε Καφέ. και έχουμε και τη συνάντηση, τη συνεδρίαση των συντονιστών. Θα έχετε και χρόνο να εργαστείτε το πάνω στο θέμα ε, που δεν θα συζητήσουμε τώρα, το Σαββατοκύριακο. Θα συζητήσουμε το θέμα της κυρίας Σάκε και οι συντονιστές σε μισή ώρα το αργότερο να είναι εδώ, γιατί θα έχουμε τελειώσει την κυρία Σάκε μέχρι τότε, οπότε θα αρχίσουμε τη συνεδρίαση των συντονιστών. Σήμερα θα μιλήσουμε για θέματα σημαντικά. Θα ήθελα, όσο περιμένουμε τη συνάδελφο, να σας προσκαλέσω τους ε, συναδέλφους ευρωβουλευτές, ε, βοηθούς, ε, συνεργάτες στο, στη μεγάλη αθλητική εκδήλωση που θα οργανώσει η Πολωνική Αντιπροσωπεία το μεγάλο το, ε, ποδοσφαιρικό γεγονός. 18 θα έχουμε εθνικές συμμετοχές, θα έχουμε και εκπροσώπους της Ισπανίας. Ε, από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ε, στην Πολωνία ε, το ποδόσφαιρο έχει πολύ βαθιές ρίζες. Μάλιστα ο κύριος Ντούντεκ που δεν θέλει και μέρος της Ρεάλ Μαδρίτης θα είναι εδώ. Πρόκειται για τεράστια αθλητική εκδήλωση γιατί πραγματικά ο αθλητισμός είναι πια κοινωτική πολιτική και χρήζει η διάζουσας προσοχής. θα ξεκινήσουν τα εγγένεια ε, με συμμετοχή του Πρόεδρου Σούλτς, της κυρίας Βασιλείου. Από τις 12 μέχρι τις 3 ε, σας προσκαλώ θερμά όλους σε αυτή την ποδοσφαιρική συνάντηση που οργανώνει η Πολωνική Αντιπροσωπεία. Δεν μπορώ δυστυχώς, είμαι στο Βεντέρ στην Κολονία για κάτι πολύ σημαντικό. Και την Τετάρτη το πρωί θα πρέπει να είμαι στην Λίντενστράσε. Ε, αυτό είναι και ένα ε, δώρο γενεθλίων. Αλλά θέλω να μου κάνουν κάτι πρωτότυπο την Τετάρτη στη Λίντενστράσε. Και θα το δείτε, στη, θα παρουσιαστώ δηλαδή ε, στη Λίντενστράσε. Δεν θα μπορέσω λοιπόν να έρθω ε, ίσως θα δω, ε, δεν θα προλάβω, θα δω το ποδόσφαιρο. Ε, ο, θα δούμε και τον κύριο ε, ε Σούλτς, είναι, θα καταφέρουμε να τον πείσουμε. Αυτό όμως είναι λίγο σεξιστικό. Τώρα, ήρθε η κυρία Σάκη, χαιρόμαστε πάρα πολύ που ήρθε και της δίνουμε μέσα στο λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και χαίρομαι ιδιαίτερες γιατί το δώρο για θελήσω σας ευθυγραμμίζεται πλήρως με το αντικείμενο αυτό της συζήτησης και αρμοδιότητα της Επιτροπής μας. Πρόκειται για κάποιες προτάσεις ε, που περιλαμβάνονται στο σχέδιο γραμμαδότης που θα δώσω στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς. Με στόχο με θέμα την ολοκλήρωση της, της ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Ένα πολύ σημαντικό θέμα για την Επιτροπή Πολιτισμού. Ελπίζω να διαβάσετε τη γνωμοδότηση είναι σύντομη, γιατί είναι γνωμοδότηση δεν είναι έκθεση. Οι προτάσεις ε, που περιλαμβάνω ε, τάσσονται υπέρ τη ενίσχυση τη υποδομή του ΤΠΕ για τη διαχείριση του ψηφιακού χάσματο. Ε, τονίζει ότι οι μικροπληρωμέ χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο με ψηφιακό τρόπο για, και έχουν πολιτιστικό περιεχόμενο. Προτείνουμε άρση των εμποδίων προκειμένου να ολοκληρωθεί η ενιαία ψηφιακή αγορά που είναι σημαντικότητα για την ανάπτυξη νόμιμων διασυνοριακών επιγραμμικών υπηρεσιών. Γιατί αυτό που ενδιαφέρει κυρίως τον κόσμο είναι το πολιτιστικό περιεχόμενο τέτοιων υπηρεσιών. Yeah, that's basically... Ε, αυτές είναι οι βασικές προτάσεις, αυτή είναι η ουσία της πρώτης, ο πυρήνας της. Θέλουμε να άρουμε τα εμπόδια στην ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε πρόσβαση σε επιγραμμικό, πολιτιστικό και καλλιτεχνικό περιεχόμενο και ελπίζω να τύχει υποστήριξη για να δώσουμε και το πρίσμα της δικής μας Επιτροπής. Δεν είναι μόνο θέμα τεχνικό, δεν είναι μόνο θέμα αγοράς και καταναλωτών, αλλά εμείς θέτουμε τους καταναλωτές και το ακροατήριο, τα ακροατήρια γενικά στο επίκεντρο της προσοχής γιατί είναι πολύ σημαντικό ο ρόλο του στο επικραμμικό περιβάλλον και λαμβάνεται υπόψη, ώστε η ενιαία ψηφιακή αγορά να βελτιώσει πραγματικά την πρόσβαση στην τέχνη, στις τέχνες και τον πολιτισμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Μάρικε. Δεν ξέρω αν λυπάμαι για όλα αυτά, όπως ε, και εσύ, γιατί ανησυχώ λίγο σε ό,τι αφορά κάποια περιεχόμενα. Πρέπει να τα μελετήσω γιατί λέει ε, ε την απασχολεί το ζήτημα της φραγής ορισμένων περιεχομένων, πράγμα που δεν ε, είναι αποτελεσματική μέθοδος. Δεν ξέρω, δεν ξέρω πώς ε, να βγάλω από τον υπολογιστή κάποια πράγματα αν δεν υπάρχει δυνατότητα φραγής. Δεν είμαι ειδική, αλλά παρακολουθώντας όλα αυτά που μπορούν να προβάλλονται χωρίς κανένα φραγμό, παιδική πορνογραφία για παράδειγμα, ναι, ε, είμαι πολύ επιφυλακτική και δεν ξέρω αν μπορώ να συμφωνήσω με όλα αυτά. Υπάρχουν όμως πολύ καλύτερα ενημερωμένοι ε, συνάδελφοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πέτρα. Ναι, αυτό είναι το σημαντικό που είπες. Νομίζω ότι καλό είναι που, είναι, που αναφέρονται αυτά στην έκθεσή σου και σε σχέση με την παιδική ε, πορνογραφία είχαμε μεγάλες αντιπαραθέσεις σε σχέση με τη φραγή, διαγραφή κλπ. Και η φραγή συνεπάγεται κινδύνους να ε, ταλαιπωρήσουμε και αθώους ή να τους συμπαρασύρουμε ε, στα μέτρα αυτά. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί λοιπόν είπαμε και αν υπάρχουν παράνομα περιεχόμενα θα πρέπει να διαγράφονται, όχι να φράσονται. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει μια διαφορά μεταξύ απάλληψης ή διαγραφής και φραγής. Και στη Γαλλία και στη Μεγάλη Βρετανία ε, είχαμε εντονότατες συζητήσεις ε, και στη Γαλλία τον νόμο και στο Ηνωμένο Βασίλειο σε σχέση με το μοντέλο που ελέγχει τις ε, ε, ροές της επικοινωνίας. Και στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας πρέπει να σταθμίσουμε πολύ προσεκτικά ατομικά δικαιώματα, το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης ε, στην πληροφορία, την ελευθερία της πληροφόρησης και τη στάθμιση του τι σημαίνει παραβίαση δικαιωμάτων του δημιουργού. Χρειάζεται μια σωστή ισορροπία λοιπόν εδώ στην προσέγγιση μας. Μην, κάνουμε, ε, μην κάψουμε τα χλωρά μαζί με τα ξερά. Είναι σωστό λοιπόν να το αναφέρουμε αυτό πάλι και να πούμε ότι υπάρχουν πολλοί που βλέπουν με κριτικό πνεύμα τους μηχανισμούς ε, φραγής σε σχέση με τα δικαιώματα του δημιουργού. Επίσης, σωστό είναι να πούμε ότι αυτό που ενδιαφέρει κυρίως είναι να έχουμε και συστήματα πληρωμής, τα οποία θα είναι απλά και εύχρηστα και η δυνατότητα ε, για νόμιμο κατέβασμα θα πρέπει να διευκολύνεται με απλό τρόπο, με νόμιμο τρόπο, ούτως ώστε να μην χρειάζεται να προσφύγει κανείς σε παράνομες σελίδες για να κατεβάσει αυτό που θέλει, επειδή είναι και ε, χαμηλό το κόστος των νόμιμων σελίδων και εύκολη η πρόσβαση σε αυτές. Αυτό είναι το σημαντικό που χρειαζόμαστε και να υπάρξει και η συνείδηση του γεγονότος ότι και η δημιουργικότητα έχει μια αξία που πρέπει να πληρώνεται. Υπ' αυτή την έννοια Νομίζω ότι η Μαριέτα Σάκε βρήκε μια καλή ισορροπία ε, και προς την κατεύθυνση της Κομισιόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Είμαι εδώ πίσω και δεν με βλέπετε. Α, μάλλον εδώ μπροστά και δεν με βλέπετε. Η έκθεση Σάκε είναι πολύ καλή και η α κάλυψε τα περισσότερα σημεία. Το θέμα των μικροπληρωμών είναι πολύ σημαντικό και ευτυχώς η, η το κάλυψε στην έκθεση της, στην γνωμοδότησή της. Αναφερθήκαμε και στο θέμα της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ψηφιοποίησης του πολιτιστικού περιεχομένου. Διαπιστώνουμε ότι ο κόσμος θέλει μουσικά έργα, θέλει βιβλία σε ψηφιακό υπόθεμα. Φυσικά θα πρέπει να διευρύνουμε το διαδίκτυο, να διαβρύνουμε την πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόμενο, να μην ξεχάσουμε και το θέμα του ραδιοφάσματος. Σημαντική η ψηφιακή Ευρώπη για μας και η ψηφιακή πολιτική θα είναι στο μέλλον από τις πιο σημαντικές από τις πιο σημαντικές. Θα πρέπει λοιπόν να επεκτείνουμε το διαδίκτυο, να διευρύνουμε την πρόσβαση, ώστε να μπορέσει ο κόσμος να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες, πλούσιες δυνατότητες που προσφέρει ο ψηφιακός κόσμος και να μπορούν να, να πραγματοποιούνται μικροπληρωμές και ε, διαδικτυακά. Είναι πολύ καλή γνωμοδότηση, δεν χρειάζεται καμία αλλαγή. Ευχαριστώ η Έμα Μακλάρκεν. Ευχαριστώ. Και εγώ επικροτώ την γνωμοδότηση ΣΑΚΕ για την ολοκλήρωση της ψηφιακής αγοράς. Εγώ είμαι ε, σκιώδη συγγήτρια και στην Επιτροπή ΙΜΚΟ και είναι αναφυσβήτητο ότι είναι τεράστιος ο οικονομικός αντίκτυπος του, διε, του διαδικτύου. 603 εκατομμύρια, 6, ε, συγγνώμη, 3 εκατομμύρια το χρόνο ε, παγκοσμίω και στην Ευρωπαϊκή Ένωση επίση ένα μεγάλο ποσό. Φυσικά το πολιτιστικό περιεχόμενο θα πρέπει να περιλαμβάνεται, αλλά να αμείβονται καλλιτέχνες για το έργο τους. Επίσης να τονίσουμε την ανάγκη προστασίας του copyright, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Επίσης το θέμα της πολυδικαιοδοσιακής άδεια είναι πολύ σημαντικό, αλλά δεν θα πρέπει να αποβεί εις βάρος της προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας. Ναι υπέρ της πρόσβασης στο ίντερνετ, αλλά όχι εις των πνευματικών δικαιωμάτων. Είναι κατακαιρματισμένα τα συστήματα δυστυχώς και υπάρχουν πολλά διαφορετικά συστήματα προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων στα διάφορα μέλη, με, κράτη-μέλη. Ε, το σύστημα iTunes είναι διαφορετικό στο ε, Ηνωμένο Βασίλειο και διαφορετικό στο Βέλγιο θα πρέπει να διευρύνουμε, να εμπλουτίσουμε την, την επιλογή που έχουν οι καταναλωτές, αλλά να προστατεύσουμε και τους δημιουργούς. Σε ό,τι αφορά τα θέματα της φραγής, θα πρέπει να έχουμε πολλά εργαλεία στη διάθεσή μας για να αναλάβουμε δράσεις. Το θέμα της πορογραφίας είναι ένα θέμα που κατ' εξοχή θα πρέπει να ασκείται το δικαίωμα αυτό της φραγής, αλλά να μην ξεχνούμε ότι θέλουμε να ολοκληρώσουμε την ενιαία ψηφιακή αγορά, να μην εμπλακούμε δηλαδή σε μια συζήτηση για ελευθερίες, διαδίκτυο, προστασία κτλ. Το δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Είμαι, είμαι, είναι θέμα ενιαίας ψηφιακής αγοράς και αυτής της βιομηχανίας υπό αυτό το πρίσμα θα πρέπει να τις καλύψουμε. Η Σαμπίνε. Και εγώ θα προσέθετα κάτι. Είναι σημαντικό το copyright και ο κατακαιρματισμός. Καλό είναι που τα αναφέρουμε και θα ήθελα όταν κάποια στιγμή υποβάλει την αναθεώρηση για το copyright κομισιόν να δει το θέμα αυτό. Καλό θα ήταν να το πούμε και στην έκθεση ε, σε σχέση με την, ε, ε, τις εταιρείε επεξεργασίας, γιατί όλα αυτά ολοκληρώνουν την ψηφιακή αγορά. Κάτι άλλο που δεν αναφέρεται είναι η βελτίωση των ευρυζωνικών δικτύων, αν θέλω να καταργήσω εμπόδια, Πρέπει να καταργήσω και τα εμπόδια στην πρόσβαση σε αυτή την αγορά. Κάποιες περιφέρειες, αγροτικές κυρίως, δεν μπορούν να αξιοποιήσουν αυτή την αγορά. Πρόκειται λοιπόν για θέλει το αποκλεισμό. Καλό θα ήταν να υπάρξει μια μνήα και αυτού. Ίσως ε, με μια τροπολογία μπορούμε να αναφερθούμε στη βελτίωση των ευρυζωνικών δικτύων ε, που ε, αναφέρεται, αναφέρονται και στην έκθεση που δεν θα συζητήσουμε σήμερα. Ε, πρέπει να διευκρινίσουμε και το λέει στην έκθεση ότι η φραγή πρέπει να είναι η ίστατη καταφυγή, όχι το πρώτο μέσον όμως πρέπει να βρούμε ενδεδειγμένες δυνατότητες ε, για να προστατεύουμε τα δικαιώματα του δημιουργού και στο διαδίκτυο. Το δικαίωμα, η ελευθερία στην πληροφορία και πρόσβαση σε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες. Κάποια στιγμή αυτό συγκρούεται με τα δικαιώματα της πνευματικής ιδιοκτησίας που πρέπει επίσης να προστατεύονται. Μπορεί να, να είναι άειλο το προϊόν, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν έχει αξία για το δημιουργό του και πρέπει να διευκρινίσουμε ότι και τα δύο δικαιώματα είναι εξίσου νόμιμα, θεμητά και πρέπει να προστατεύονται. Και πρέπει να ενισχύσουμε τις δυνατότητες εξέβρασης νόμιμων μέσων για την προστασία. Όσο περισσότερα νόμιμα μέσα διαθέτουμε, τόσο λιγότερο θα χρειάζεται να προσφεύγει κανείς σε παράνομες πλατφόρμες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως και οι προλαλήσαντες συμφωνώ το άρθρο 7 είναι πάρα πολύ σημαντικό, η παράγραφος 7 μάλλον, και το γεγονός ότι ε, επιβάλλουμε κυρώσεις ή φράσουμε δεν είναι καλή πρόταση. Είχαμε ε, και σε επίπεδο την άκτα και σε επίπεδο γαλλικό μια σύμβαση για την πνευματική ιδιοκτησία. Νομίζω ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη πρόσβαση των πολιτών στο πολιτιστικό περιεχόμενο. Νομίζω ότι με το καταποκοπή ποσό θα μπορούσαμε να έχουμε ε, πρόσβαση σε ένα πολύ πλούσιο περιεχόμενο που είναι πολύ σημαντικό. Συμφωνώ με την πρόταση της ε, για το γεγονός ότι ε, η δυνατότητα φραγής, η, αυτή η κύρωση της δυνατότητας φραγής χρησιμοποιήθηκε κατεξοχήν από αυταρχικά καθεστώτα, της Τινησίας, της Κίνας. Είναι σημαντικό λοιπόν να μην προβλέψουμε αυτή τη δυνατότητα αυταρχικής φραγής, ανεξέλεγκτης, γιατί μην ξεχνάμε ότι η πρόσβαση στο Ιντερνετ είναι θέμα ελευθερίας των πολιτών. Οι πολίτες είναι ελεύθεροι να εξετάσουν οποιοδήποτε πολιτιστικό περιεχόμενο θέλουν. Ναι, αλλά εδώ μιλάμε για την εσωτερική αγορά, όχι για την Κίνα ή κάποιο καταπιεστικό καθεστώς. Μιλάμε για την εσωτερική αγορά μας. Και νομίζω ότι μπορούμε να ε, εστιάσουμε περισσότερο στα δικά μας εδώ. Το θέμα copyright βέβαια, το οποίο πάντοτε ανακύπτει στη συζήτηση για τα μέσα, δεν μπορεί εδώ να υποβαθμιστεί. Αν δεν έχουμε δημιουργούς, δεν θα ε, έχουμε και όφελος. Στο σημείο 4 λοιπόν, όσοι από την ομάδα μου ε, θέλουν μπορούν ε, ίσως να σκεφτούν να, να καταθέσουν μια τροπολογία. Επίσης, ε, αν αφήσουμε το 7 ως έχει, θα αφήσουμε το 7 ως έχει ή θα κάνουμε μια πρόταση και αναφερόμενη στο θέμα της παιδικής πορνογραφίας να μην υπάρχει φραγή αλλά διαγραφή Ίσως μπορούμε και εκεί να πούμε κάτι. Το είπε και η κυρία Κάμερε Φέρτε. Ο κύριος Μπόρις ζητεί το λόγο τώρα. Αν μιλούμε για ενιαία ολοκληρωμένη ψηφιακή αγορά, θα πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα τον αποκλεισμό πολλών συμπολιτών μας από την πρόσβαση στο ίντερνετ. Θα πρέπει λοιπόν να καταπολεμήσουμε αυτόν τον ψηφιακό αποκλεισμό που βιώνουν πολλοί συμπολίτε και να ταχθούμε υπέρ του ψηφιακού αλφαβητισμού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό μήνυμα. Εκτός από την έλλειψη πρόσβασης στο ίντερνετ για πολλούς πολίτες, έχουμε και κάποια νομικά εμπόδια, κάποια νομικά κολλήματα. Καλό θα ήταν να εναρμονίσουμε ή να ενοποιήσουμε και τα νομικά καθεστώτα που ισχύουν για το ίντερνετ. Είναι σκανδαλώδες το γεγονός ότι εκπρόσωποι πολλών χωρών μελών δεν μπορούν να ε, πραγματοποιήσουν ε, ε, πληρωμές online, γιατί δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις πιστοτικές τους κάρτες σε όλα τα κράτη-μέλη. Είναι πολύ σημαντικό νομικό κόλλημα αυτό. Θα μπορούσαμε λοιπόν να απαιτήσουμε κάποιες δράσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή να έχουμε πανευρωπαϊκές άδειες. Άλλωστε προς αυτήν την κατεύθυνση βαίνουμε. Και είναι σημαντικά τα θέματα, τα οπτικοακουστικά και τα μουσικά. Ε, εκεί προσπαθούμε να βάλουμε μια εναρμόνιση, αλλά μπορούσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαιτήσουμε πολύ τολμηρές προτάσεις για κάποια νέα μοντέλα λειτουργίας της ψηφιακής αγοράς. Δεν ξέρω αν θα έχουμε ένα σύστημα αποκόπη πληρωμής ή να πληρώνουμε με, ε, τα πνευματικά δικαιώματα με κάθε κλικ που κάνουμε θα πρέπει να υπάρχει μια εναρμόνιση ότι αφορά τη δυνατότητα αγορά ψηφιακού περιεχομένου, γιατί δεν υποβάλλει ε, ούτε επιχειρησιακά μοντέλα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτε διάφορε νομικέ επιλογέ δεν προτείνει. Ο ψηφιακό κόσμο εκτιλήσεται ραγδαία. Οι νέοι απαιτούν από εμά μεγαλύτερη δραστηριοποίηση και μεγαλύτερη τόλμη. Παρακαλώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επευκαιρία αυτή τη να αξιοποιήσει τις ε, συστάσεις και να υποβάλει πολύ τολμηρές προτάσεις για νέα μοντέλα και νέα εναρμόνιση. Ευχαριστώ. Λοιπόν, διαπιστώνω ξανά ότι δεν υπάρχει κανείς από την Κομισιόν. Εν τω μεταξύ ήρθε κάποιος υπεύθυνο για τα προηγούμενα θέματα. Έφυγε όμως εν τω μεταξύ. Αυτό είναι πολύ δυσάρεστο. Κάποιος ε, δεν μπορούσε να έρθει γιατί ήταν στην ε, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή που δεν μπόρεσε να έρθει σε εμάς. Τώρα δεν υπάρχει κανείς. Αξιοσημείωτο και απαράδεκτο. Εγώ θα ενημερώσω την Επίτροπο και γραπτός. Εσείς είστε πάντα εδώ, αλλά δεν μπορείτε να αντικαταστήσετε αυτούς που πρέπει. Ξέρω ότι στενοχωριέστε κι εσείς και είστε πολύ εντάξει. Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη για την κατάσταση που προέκυψε ο αρμόδιος είχε έρθει για το σημείο 8. Θα ξαναέρθει σήμερα το απόγευμα στο τέλος της συνεδρίασης. Οι συνάδελφοι τώρα της ε, Γενικής Διάθεσης ΕΦΣΟ είχαν ειδοποιηθεί ότι το σημείο τους θα συζητιόταν στις 10 η ώρα. Ήρθαν πολύ αργά, ε, δεν έφταγαν εκείνοι, τους είχαν πει 10. Γενικώ πώς σας παρακολουθούμε εμείς από πλευράς Κομισιόν, εσάς στην Επιτροπή Πολιτισμού και είναι η πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό που, δεν είχαμε, που είχαμε όλα αυτά τα προβλήματα. Ε, ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι δουλεύουν παράλληλα πολλές επιτροπές. Ζητούμε συγγνώμη γι' αυτό, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να παρακολουθούμε τις εργασίες σας. Also, Δεν το πιστεύω ότι κάνετε ό,τι μπορείτε για να μας βοηθήσετε. Εσείς ναι, αλλά όχι η Κομισιόν και το ξαναλέω. Έτσι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Όταν είναι στην ημερήσια διάταξη πρέπει να είναι κανείς εκεί. Ίσως όχι από τις 9, αλλά δεν πρέπει να υποθέτει κανείς ότι η ημερήσια διάταξη θα ε, ισχύει ως έχει, μπορεί να αλλάζει ανά πάσα στιγμή. Σήμερα μπορεί να κάνουμε αλλαγές. Πρέπει λοιπόν να ε, τους ενημερώνετε ότι πρέπει να έρθουν. Μπορεί να μην μπορούσατε να τους βρείτε. Εν πάση περιπτώσει εσείς κάνετε ό,τι μπορείτε πρέπει να σεβόμαστε τα θεσμικά όργανα. Εμείς στην Κομισιόν τη σεβόμαστε, να σέβεται και εκείνη το Κοινοβούλιο. Θα γράψουμε λοιπόν μία ε, φιλική, ε, λιγότερο φιλική επιστολή και θα τα πούμε όλα αυτά. Η Μαρίκε. Μαριέτα. Σύντομα. Χαίρομαι για τα σχόλιά σας. Υπάρχει ευρεία συνένεση νομίζω για την ανάγκη να αυξήσουμε το νομικό περιεχόμενο που υπάρχει διαθέσιμο μέσω εύκολης ε, πληρωμής αλλά και μέσω τολμηρών προτάσεων, όπως είπε ο συνάδελφος, ε, για εναρμόνιση, για μεταρρύθμιση ή, εν πάση για πιο εύκολες μορφές ε, copyright και πιο εύκολο διαχειρίσιμο copyright. η πρόταση για διαγραφή αντί για φραγή ιστοσελίδων είναι μια πρόταση που την κρατάω. Είναι πολύ σημαντικό να διακρίνουμε ότι δεν μιλάμε για εγκλήματα όπως η παιδική πορνογραφία. Αναμφίβολα, αυτά είναι τα χειρότερα πιθανά εγκλήματα. Μιλάμε για κάποια πράγματα ε, όμορφα που είναι το πολιτιστικό περιεχόμενο επιγραμμικά. Ε, κάτι που ενδιαφέρει τον κόσμο. Υπάρχουν πολλές σχολές σκέψης. Ορισμένοι μιλάνε για την εφαρμογή, άλλοι μιλάνε για το περισσότερες ευκαιρίες. Το θέμα είναι αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες της ψηφιακής αγοράς, όπως ανέφερε και η συνάδελφος που ασχολείται με θέματα εσωτερικής αγοράς. Εμείς ως Επιτροπή μπορούμε να εστιάσουμε στην αύξηση του νομικού περιεχομένου ως αντίβαρο για τη ζήτηση παράνομου περιεχομένου, νόμιμου περιεχομένου, συγγνώμη. Ε, με αυτόν τον τρόπο θα γλιτώσουμε και δημόσια κονδύλια Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την εφαρμογή. Ξαναλέω ότι εκτιμώ όλα σας τα σχόλια. Μπορείτε να ζητήσετε περισσότερες διευκρινήσεις μέσω συστάσεων και μπορούμε να κάνουμε μια καλή... μέσω τροπολογιών, και μπορούμε να κάνουμε καλές συστάσεις στην Επιτροπή και ελπίζω να μας ακούσουν και μέσα στο Κοινοβούλιο αλλά και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Στις 5 Ιουνίου, όχι, Α, 5 Ιουνίου, ναι. Ε, 12 το μεσημέρι, προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών για την πρόταση της Μαράικε. Κάποιοι συναδελφοί μίλησαν για την διαγραφή, τα ευρεζονικά ε, ε, και κάποια άλλα θέματα ακόμη. Ας καταθέσουν τροπολογίες και στην επόμενη συνεδρίαση θα αποφασίσουμε και επί αυτών των τροπολογιών για να μην τα αναλάβει η Μαράικε. Η έκθεση Φοντάνα θα συζητηθεί το απόγευμα. Ε, λύεται η συνεδρίαση. Παρακαλώ τους συναδέλφους συντονιστές να παραμείνουν γιατί έχουμε μια πολύ σημαντική συνεδρίαση με κάποιες αποφάσεις που πρέπει να λάβουμε.